Κυρίε uh, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα προεδρεύσω με πολύ ηρεμία. Κανονικά έπρεπε να είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω πρόβλημα στο λαιμό μου, στην τραχεία μου, στο θώρακά μου, αλλά Είμαι εδώ. Είμαι εδώ γιατί προετοιμαζόμουν επί έξι μήνες ψυχολογικά για να είμαι σε αυτή την ψηφοφορία. Ήταν αδύνατο να τη χάσω λοιπόν. Ήσυχη θέλω να είναι η ψηφοφορία γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Ορισμένες, ε, ορισμένες συμβαστικές τροπολογίες θα περάσουν είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση βραχία κεφαλή και θα είναι δύσκολο. Ε, και έχουμε χρόνο μέχρι τις 12.30. Επομένως, ας προχωρήσουμε βαθμιδών και μπορεί να χρειαστεί και ένα πεντάλεπτο διάλειμμα κάπου στα μισά ε, για λόγους υγείας, για μένα το, θα το κάνω, έτσι. Ήθελα να σας τα πω αυτά προκαταρτικά. Και τώρα, πάμε να τσεκάρουμε για την α, ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Λειτουργεί. Κλείνω την ψηφοφορία. Ε, ξεκάθαρη απάντηση. Όλοι έχουν αισιοδοξία από ό,τι βλέπω. Πάμε στην πρόταση για οδηγία. Διορθώνω. Στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Κάρτας Υπηρεσιών και Συναφών Διοικητικών Διευκολύσεων. Η συντάκτη είναι η κυρία Μαρία Σπυράκη. Τέσσερις τροπολογίες που είναι πανομοιότυπες. Θα τις ψηφίσουμε και μάλιστα ηλεκτρονικά από την αρχή παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Και τις τέσσερις τροπολογίες ομού. Άρχεται ψηφοφορία. Ε, one SND too Ένας υπεράριθμος σοσιαλιστής ψηφίζει. One SND. Now is okay. Εντάξει τώρα, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αγαπητοί φίλοι, τι σημαίνει η απόφασή μας. Σημαίνει και θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Απορρίπτουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει η απόφασή μας. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Οπότε αν θέλουμε να δεχτούμε την απόρριψη της πρότασης, θα πρέπει στην τελική ονομαστική ψηφοφορία να ψηφίσουμε ναι. Δηλαδή ναι στην απόρριψη. Αν τώρα πούμε όχι, σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώμη. Υπάρχει πολιτική διαφορά μεταξύ των δύο στάσεων. Αν πούμε απόρριψη θα πρέπει να ψηφίσουμε ναι. Αν ψηφίσουμε όχι είναι σαν να μην δίνουμε καμία γνώμη. Τελική ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. And I close the vote. γίνεται δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίσαμε την απόρριψη. Η γνωμοδότησή μας είναι απλή. Απορρίπτουμε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν το της. Πάμε τώρα στη δεύτερη έκθεση της κυρίας Πυράκη, που είναι μια οδηγία για το ίδιο θέμα. Τέσσερις τροπολογίες έχουμε στην αρχή Τις ψηφίζουμε μαζί. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Αυτό σημαίνει το ίδιο πράγμα. Απόρριψη. Στην τελική ψηφοφορία, αν ψηφίσουμε ναι, είναι απόρριψη. Αν δεν υπάρχει ξεκνομοδότηση, σημαίνει ότι έχουμε ψηφίσει όχι. Αποδεκτό. Απορρίψαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα πάμε στην έκθεση του Χωσέ Μπλάνκο Λόπεθ. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Συμβασμός 1α. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είναι Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός αναμπή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφοφορίας. Έχουμε έναν από το άλλο παραπάνω. Εντάξει τώρα πέρα σφοφορία. Δεκτό. Τώρα πάμε στη σελίδα 14. Τροπολογία 22. Σας δίνω χρόνο να βρείτε την τροπολογία 22. Στη δική μου σελίδα υπαριθμό 14. Δεν έχουμε κατά το ίδιο κείμενο. Πάνω κάτω στη 14 θα τη βρείτε. Τροπολογία 22. υπέρ, κατά, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 22. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 81. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αποδεκτή. Τελικά πρέπει να ελέγχουμε κάθε τροπολογία. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. Προχωράμε. Πηδάμε δύο σελίδες. 369. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 370. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε χρονικά 370. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τρεις ίδιες τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. 418 μέχρι 84. Ζητώ συγγνώμη. 381. Υπέρ. Διαφωνεί ο Κατά. Ελέγχουμε την 381. Πέρας φοφορίας Απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρεις τροπολογίες. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 418 μέχρι 34 421 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 431 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πάμε στην επόμενη σελίδα. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 453. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρεις ίδιες τροπολογίες. Από την 464 μέχρι την 455. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 39. Υπέρ. Κατά. Ας την ελέγξουμε. Την 39. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 468 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 468. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω έτσι. Ποιοι είστε υπέρ, ποιοι είστε κατά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε 468. Απορρίπτεται. 457 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 456 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 456. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 460 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 462 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 466 υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την 466 ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 465 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά, αποχές, δεκτός. Πάμε τώρα στη σελίδα 27, 88. Υπέρ, κατά. Δεν σηκώνει τα χέρια σας, πρέπει να τα ελέγξουμε ευθονικά. Ψηφίζουμε την 88. Πέρας φοφορίας. Δεκτή. 608 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το συμβασμό, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Συμβασμός 4. Πέρας φοφορίας δεκτός. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές δεκτός. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτός. Τροπολογία 687 υπέρ με τις τρεις υπόλοιπες. Τέσσερις τροπολογίες. από την 687 μέχρι την 852 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 691 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 694 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τρεις τροπολογίες μαγής, από την 23 μέχρι την 25 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 696 υπέρ, κατά, την ελέγχουμε. 696. Απορρίπτεται. 703 και 50 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο τροπολογίες. 793 και 106 υπέρ κατά. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ αυτές τις δύο τροπολογίες. Πέρας τους οφορίες. απορρίπτονται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 682 και 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 814 ε, υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 814. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 8 50 και 59 υπέρ, κατά, αποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της φοφορίας Απορρίπτονται. Και 8-16 υπέρ, κατά. Να ξαναψηφίσουμε να το ελέγξουμε και αυτό. 8-16. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίπτεται. 8, 18 και 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και πάμε στην 817, πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Να ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 817, στους οφορίες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Και πάμε στην 820. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 820. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 10 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 μαζί με προφορική τροπολογία. Κατά, είναι κανείς κατά. Δεν καταψηφίζει κανείς, δεν διαφωνεί κανείς, οπότε μπορούμε μάλλον να ψηφίσουμε, όπως είχαμε συμφωνήσει. Συμβαστική 11, υπέρ, κατά. Να ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά είναι σημαντική αυτή η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε επί της ε, συμβαστικής τροπολογίας 11 με προφορική τροπολογία πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 877 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 878 μαζί με την 879 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται επίσης. Ψηφίσαμε για δύο τροπολογίες, την 78 και την 79. 880 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάμε στην 898 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε. Για την τροπολογία 898 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 899 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 900 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 904 ε, υπέρ κατά, αποχές. Δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας. 904. Vote 901, sorry, this wrong. We have to vote this. Ah. Because this is, was not adopted. Eh, moment, moment, dear friends. Μια στιγμή. Παρατήρηση της γραμματείας είναι πολύ σημαντική. Δεν εγκρίθηκε η 899 που σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 901. Είναι μεγάλη διαφορά αυτή γιατί δεν έγινε δεκτή η τροπολογία 899. Δεν υπερψηφίστηκε, δεν εγκρίθηκε. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία για την τροπολογία 901, υπέρ.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 901. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και γι' αυτό πάμε αργά-αργά. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά δυστυχώς πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 901. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 904. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 904. Πέρας. Η 902 υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. I close the vote. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 9-12. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Μαζί με την 9-13. 9-12, 9-13. Ψηφίζουμε από κοινού. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 914. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε 10 σελίδες μετά, συμβαστική 13, στη δική μου σελίδα 62, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ, μαζί με προφορική τροπολογία σε αυτήν που την χάνει τη στήριξη όλων των ομάδων η προφορική τροπολογία. Λοιπόν, συμβαστική 15 μαζί με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας, συμβαστικής τροπολογίας 17, πάρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ για τη συμβαστική 17, πέρας ψηφοφορίας. Με τεράστια πλειοψηφία υπερψηφίζεται, εγκρίνεται. Και πάμε στην 126-127. Ε, Υπέρ 1267, συγγνώμη. Περιμένω, περιμένω. Στη δική μου σελίδα 94, 94-1267, Υπέρ, κατάποχες απορρίπτεται. Πάμε 1268 και 1269 υπέρ μαζί κατά να το ελέγξουμε. Πέρα στις οφορίες εγκρίνονται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά Εποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές. I εβδομήντα. No. No. 1270. Uh, υπέρ. Κατά. Αποχές. 40 uh, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1277 υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα, για την τροπολογία 1277 στις ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική 19, τρεις σελίδες παρακάτω. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 28. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρος. Ξανά. Σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ για την τροπολογία. 29 ψηφίζουμε. 29. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 6. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Συνάδελφοι από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας, ψηφίζετε κανονικά. Τρυπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Sorry for your work, hard work. Λυπάμαι που σας κουράζω. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. Τέλος ψηφοφορίας. Οι δύο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία. I close Accepted. Τέλος ε, ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το έλεγχο δεν ψηφίζει καν. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 11 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 πάλι, αλλά της Επιτροπής έμβει αυτή τη φορά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της έμβει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 178 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας υπεράριθμος από το ΕΛΚ ψηφίζει. Δεν πειράζει γιατί τους ή είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται 194. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Επαναλαμβάνω. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 194. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 177. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν ψηφίζουν οι βουλευτές. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μάλλον και άλλοι είναι για το νοσοκομείο. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Τζανονάτο Μάλλον λάθος έγινε. 192 έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται ψηφοφορία. Καλή πρόταση για ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στις τροπολογίες 193 και 14 μαζί. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Άποχες. Απορρίπτονται. 195 και 15 μαζί. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 και 20 μαζί υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 207 και 20 άρχιτη ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτονται 210 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 213 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 214. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 214. Τροπολογία 215 Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 11 και 22 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 11 και 22 τροπολογίες. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 216. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Και πάλι χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη 216 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την 23. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 218 και 219, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες 218 και 219. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνονται με εμφανή διαφορά. Τροπολογίες 244 και 245. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικό έλεγχος για τις τροπολογίες 244 και 245. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Τώρα, τροπολογίες 241, 242 και 243 μαζί, υπέρ, κατά, Θεούλη μου, Ηλεκτρονικό έλεγχος και πάλι χρειάζεται. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Έχουμε άλλες τρεις τροπολογίες, 2.46, 2.47 και 2.48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές και πάλι ηλεκτρονική επαλήθευση χρειάζεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Τέλος. Απορρίπτονται. 254. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.55 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.55 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 256 και 257 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία για την 259 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 260 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται, δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 260, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 261 άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. Rejected. Απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και πάλι για τη 262 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τέλειο αποτέλεσμα. Φανταστικό. Παναγίτσα μου. 2,64 υπέρ. Κατά. Τώρα μάλλον ισοπαλία θα είναι. Πολύ κοντά τέλο πάντων. 2,64 άρχεται η ψηφοφορία. Είπαμε ισοπαλία. Καλό να το ελέγξουμε λοιπόν. 2,64 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.70 γυρνάμε σελίδα. 2.70 γυρνάμε σελίδα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για 270 άρχεται η ψηφοφορία. Accepted. Accepted. 271. 271 γιατί 270 εγκρίθηκε, 270 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 18. Τέλος. Απορρίπτεται. 19 και 2,72 μαζί υπέρ. Κατά. Χρειάζεται και για αυτές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 19 και την 272. Rejected. Two... Απορρίπτονται. 2,73 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 273. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 274 υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. 274. 274. Ηλεκτρονικός έλεγχος, μια και το ζητάτε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 278. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 278. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 277. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 279. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 282. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ασαφές το αποτέλεσμα. 285. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. 282, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας, συντριπτική πλειοψηφία. Ε, λαμπρό αποτέλεσμα. Τέτοιος έλεγχος δεν έχει ξαναγίνει. Άνευ προηγουμένου επιτυχία. Επόμενη σελίδα 285. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.87 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 2.87 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία για την 288. Accepted. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ηλεκτρονικός έλεγχο και για την 22. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ε, 290 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 291 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 291 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 33 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 33 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τριακόσια υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρεις τροπολογίες τώρα. 318, 319 και 42. Πανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 320 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 320. Άρχεται ψηφοφορία. I close the vote. Τέλος. Απορρίπτεται. 54. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. ΔΕΒ 16. Πάμε επόμενη σελίδα και στην τροπολογία 16 της ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 16 της ΔΕΒΕ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 18 της ΔΕΒΕ. And I close the Accepted. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 93. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 93... Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται... Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίθηκε λοιπόν η έκθεσή μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, εισηγητές και οδησηγητές στη γραμματεία, ε, της γραμματείας των πολιτικών ομάδων και της δικής μου φυσικά, για την προσπάθεια που κάναμε, για τις εργασίες μας που συνεχίζονται γιατί ακούγοντας τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και αυτές που προωθούν κάποια κράτη-μέλη ε, διαπιστώνουμε ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο, έχουν ανάψει όλα τα καμπανάκια. Πάντως ε, με τη θέση αυτή ε, επιδεικνύουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία για την υλοποίηση των στόχων του Παρισιού. Και χάρη στην έκθεση αυτή προωθούμε μια οδηγία που πραγματικά θα συνάδει με τις συμφωνίες του Παρισιού για το περιβάλλον. Νομίζω ότι ήταν πολύ αίσια η διεξαγωγή και η έκβαση της ψηφοφορίας. Ελπίζω να ενισχυθεί με το αποτέλεσμα στην Ολομέλεια, γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε για μια ενεργειακή μετάβαση που θα μας οδηγήσει σε μια καθαρή ενέργεια. Ευχαριστώ. Στο συναδελφοί και για, τον, για την αισιόδοξη στάση σας. Ελπίζουμε ότι όλες οι χώρες ανά τον κόσμο θα ακολουθήσουν την ίδια τραπό. Και τώρα θα ήθελα να πιω κάτι στην υγειά σας, αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό διάλειμμα. Μην φύγετε από τις θέσεις σας. Καθίστε παρακαλώ εκεί που είστε. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill case. Ε, εδώ έχει πολύ περισσότερο ενόπνευμα από στην περίπτωση του, από ό,τι είχε ο Τσόρτσιλ στο δικό του ποτό. Reinhold, we vote immediately. We vote. Okay. Dear colleagues, One minute past. Πέρασε το ένα λεπτό, συνάδελφοι. Και περνάμε στο σχέδιο έκθεσης για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Όπως βλέπετε, σήμερα δεν είμαι και τόσο αποδοτικός εγώ. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την ηλεκτρονική ψήφο, ψηφοφορία του συμβασμού 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το συμβασμό 1. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Κρίνεται. Τώρα περνάμε στο mv 21. Σημείο 2. Υπέρ. Το βρήκατε. mv 21. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας φοβορίας. Δεκτή. Πάμε τώρα σε δύο τροπολογίες. 2.48 και 2.49. Δεύτερο τμήμα και στις δύο περιπτώσεις. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 2.68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Την ελέγχουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ή 34. 2,69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε χρονικά τη 2,72. Πέρας ψηφοφορίας. αποδεκτή. 40 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε χρονικά τη 40. Μία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τέσσερις τροπολογίες. Από τη 42 μέχρι την 79 στον κατάλογο. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τις ελέγχουμε. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτονται. 43. Μέχρι 31. Μέχρι 31. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτονται. 45. Και 2,78. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν σηκώνετε τα χέρια. Ψηφίσουμε τη 45 και την 278 ηλεκτρονικά ξανά. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Σας παρακαλώ. Σηκώντε τα χέρια σας. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ξανά τη 46 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 δι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα, τρεις, έξι τροπολογίες. Όχι, δέκα τροπολογίες. Έντεκα μάλλον. Στην επόμενη σελίδα. Από τη 267 μέχρι τη 285 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτός. Και τώρα πάμε 4-5 σελίδες μετά στην τροπολογία, στις δεξίες 341 και 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 343 υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 343. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε το συμβασμό 3. Σημαντικό θέμα, ο συμβασμός υπαριθμών 3. Πέρας προφορίας. Δεκτός. Συμβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Την ελέγχουμε αυτή την τροπολογία, γιατί είμαστε διαιρεμένοι σε αυτόν τον πολύ σημαντικό συμβιβασμό. Ψηφίζουμε τον συμβασμό 4. Πέρας προφορίας. Δεκτός. Είναι ανταγωνιστικές αυτές οι δύο τροπολογίες, ο 4 και ο 4α. Πάμε στην 15 στη δική μου σελίδα 31. Στην 482. Υπέρ. Υπέρ της 482 κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 5 ε, υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτός. 6 υπέρ. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτός. 486, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κάτα. Αποχές. Πρέπει να την ελέγξουμε. Πέραση φορείας. Ω Θεέ μου. Απορρίπτεται. Βλέπετε, απορρίφθηκε. 492 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 492. Θα πρέπει να σα αντιμετωπίσουμε το δύο τρόπο, κυρία Αντιπρόεδρε, με εσά, αλλά θα πρέπει να σα καταψηφίσουν και εσά οι συνάδελφοι. Πέρα τη φοφορία. Ω Θεέ μου! Εσεί κερδίσατε! 4,93 και 4,94. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. 4,95D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 496 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Οι σοσιαλιστές όμως δεν συνεργάζονται. Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν ψηφίζουν. Συμβασμός 7 είναι ο επόμενος που ανταγωνίζεται τον συμβασμό 7α. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Το συμβασμό 7 καταρχήν. Πέρας προφορίας. Δεκτός. Πάμε τώρα μερικές σελίδες μπροστά. 4.98. βρέστε την. Με ηρεμία. Σας περιμένω. 4.98 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έμβη 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την έμβη 33 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 510 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε εκτονικά την 510. Πέρας φοβορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚΑ ψήφισε. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 511 υπέρ. Κατά. Πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά και αυτήν. Την 511 δηλαδή. Πέρα της 50. Ε, θαυμάσιο αποτέλεσμα. 512 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το 512. Πέρα σχοφορίας. Απορρίπτεται. 513 υπέρ. Κατά. Χ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 513. Πέρα σχοφορίας. Απορρίπτεται. 514 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 515 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 516 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 517 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 518 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 519 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 521 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 522 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 523 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε χρονικά την 523. Πέρας πληροφορίας. Δεκτή. 524 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 500, 534 D Όχι, 524 πρώτα. Ελέγχουμε την 524. περας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Δεκτή. 534D υπέρ. Μαζί με την 535D και τις δύο. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τις δύο αυτές τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 537 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 538. Με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Γιατί ψηφίσαμε ναι στο πρώτο. Ψηφίζουμε λοιπόν και το δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Πέρας φοφορίας. Δεκτή. Δεκτό και αυτό. Και τώρα πάμε στην 539. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 539. Πέρας Απορρίπτεται. 540 υπέρ. Κατά. Αποχές. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν. 540. Πέρα φορίες. Απορρίπτεται. 542 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 543 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε. 543. Πέρα της Απορρίπτεται. Έχουμε χρόνο. MV35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την MV35. And we close the vote. Της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να την ελέγξουμε. Πέρας για την MV36 απορρίπτεται. Και τώρα τρεις τροπολογίες μαζί. 544D μέχρι την 548D. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 546 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 546. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Πάμε στην 549. 549 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία αυτή, 549. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 550 υπέρ. Κατά. εποχές δεκτή. 551 υπέρ. Κατά. εποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 551. Πέρας ψηφοφορίας. 551. Δεκτή 551. Συμβιβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτός. Πηδάμε λίγες σελίδες. 592D. Τη βρήκατε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 593 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε στην 595, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 613D, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 614, υπέρ. Κατά, να ελέγξουμε. 6-14 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφοριες εγκρινεται Εγκρίνεται. 6-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6-18 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 618, 18 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 44 ένβη υπέρ. Κατά. Ποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Να είμαστε σίγουροι. Έχουμε λίγο χρόνο έτσι κι αλλιώς. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 619 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε για την, για την 619 παρακαλώ. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται. 621 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ας ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε για την 621. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες μαζί. 623-624. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Αμφότερες. 625 υπέρ κατά αποχές ε, Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τέσσερις σελίδες και πάμε στην NV45 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. NV45. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Και πάμε στην 634-635. Υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ επί των δύο αυτών τροπολογιών, πέρας της Απορρίπτονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε δύο ανταγωνιστικές τροπολογίες, 11 και 11α. Για την ε, τροπολογία 11 ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με όχι πολύ μεγάλη διαφορά. 11 αλφα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση της προφορίες. Εγκρίνεται. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε τέσσερις σελίδες παρακάτω. Συμβαστική 11β. Υπέρ. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να είμαστε σίγουροι. Συμβαστική 11β. Ψηφίστε παρακαλώ. Καλύτερα να, να ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Τέσσερις σελίδες παρακάτω. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6.93 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ επί της 6.93. 6.93, πέρασε. Ένας υπεραριθμός από το ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει, πέρας, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρεις σελίδες παρακάτω. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά δεν ξέρω δεν είμαι σίγουρος 101 καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να είμαστε σίγουροι Πέρας. Απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά εγκρίνεται επίσης. Οπότε περνάμε στην 138 και την 139 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ευχαριστώ Πατρίτσια. Με τη βοήθειά σου τα καταφέρνω όλα. 141 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, απο... ας ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για να το επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ επί της 143, τροπολογία 143, ψηφίστε. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 142. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Compromise 17. Electronic Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της 17. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. εγκρίνεται. 7 και 151 από κοινού υπέρ, κατά, καλύτερα να το ελέγξουμε. Δύο τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Επόμενη σελίδα. Δύο τροπολογίες ψηφίζουμε. 162 και 163. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 175. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, καλύτερα να το ελέγξουμε να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 182. Επίσης κατά τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να το ελέγξουμε καλύτερα το δεύτερο τμήμα Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε καλύτερα. Για την 183 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. NV11 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, σας παρακαλώ, για την 198 τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά καλύτερα να το ελέγξουμε να είμαστε σίγουροι ψηφίστε παρακαλώ Συμβαστική 19 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.17 υπέρ, κατά, αποχές. Split vote. Part one. In favor. Κατά τμήματα. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά 225 να ψηφίσουμε ευχαρίστως. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας σοφορίας. Απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.29 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε. 2.29, 2.29, ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά, επί της τροπολογίας 2.29, πέρας, απορρίπτεται. 2.38 υπέρ, 2.30 υπέρ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.44 υπέρ κατά να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της 2.44. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.45 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε καλύτερα. 83. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Και 84 υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 84, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση Κομισιόν, όπως έχει τροποποιηθεί. Με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Uh, uh, Αντιλαμβάνομαι ότι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι, δεν έχω αρκετή ενέργεια για σας σήμερα. Να σας υπενθυμίσω το ραντεβού μας στις 2.30. Θα ξαναρχίσουμε στις 2.30. Έχετε τρεις ώρες ελεύθερο χρόνο. Χάρη στην καλή μας οργάνωση τελειώσαμε νωρίτερα. Ευχαριστώ και ραντεβού στις 2.30.